16. Κοινό ψήφισμα τριών πολιτικών, τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Αρχίζω με την 40, με τη, στην παράγραφο 1, νομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία για το τμήμα πρώτο. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο, με τα ανέγερση χειρών, με χειρών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 με ανάταση χειρών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρο. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 για την παράγραφο 4 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 4 σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία για το υπαριθμόν 2 τμήμα. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτό το τμήμα Τροπολογία μόνο 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία μόνο 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 6. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σκοπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 7 αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα πρώτο ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει πέρας Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 11, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 13, σε δύο τμήματα, πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τέλος απορρίπτεται τροπολογία 12 ονομαστική αρχίζει τέλος απορρίπτεται. 13 ονομαστική ψηφοφορία πάντα αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 9 ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 Επίσης ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 16 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. δύο Ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπάρχει μόνο 10, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας.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 Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει όμως τότε η υπαριθμόν 27. Ψηφίζουμε την παράγραφο 20 στο αρχικό κείμενο. Α, όχι, μια στιγμή. Και αυτή η εκπίπτει λοιπόν. Ωραία. Επιταχύνουμε τότε. Παράγραφος 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο σε ονομαστική ψηφοφορία, η οποία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο. Υπέρ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 αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται παράγραφος 30, 31 ονομαστικά αρχίζει πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 32 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 33 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 6 ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και άρα δεν απαιτείται να ψηφιστεί το αρχικό κείμενο. Τροπολογία 29 των φιλελευθέρων ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τώρα σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει. Τέλος, εγκρίνεται. Τμήμα τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ, Θέλετε να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία του τμήματος 3 της 35. Ε, ηλεκτρονικά αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήταν σαφέστατο το αποτέλεσμα. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα, τις 36 λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα τρίτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 37. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομοίως. Για το αρχικό κείμενο της 39 ζητείται ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές, Ομοίως εγκρίνεται. 43 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και αυτό Τροπολογία υπαριθμών 4 των πρασίνων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 31. 31 των φιλελευθέρων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ομοίως. Αρχικό κείμενο της 47 πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό το τμήμα. παράφορ 48. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση του δευτέρου τμήματος. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Ονομαστική τώρα για το τρίτο τμήμα. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τμήμα τέταρτο. Επίσης ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 55. Αρχικό κείμενο. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα αρχίζει. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 56 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 57. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της 58, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 60. Αρχικό κείμενο, πέντε τμήματα. Πρώτο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα πέμπτο ονομαστικά και πάλι αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 61. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 37 των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Α, ευχαρίστως να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 37. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται και ζητώ συγγνώμη. Παράγραφος 63. Αρχικό κείμενο. Τέσσερα τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Τρία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 65 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 τμήμα δεύτερο συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό Παράγραφος 67, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 70, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 72, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 των Σοσιαλδημοκρατών. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι ορισμένοι δεν συμμετέσχουν καν στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να επαναληφθεί υπέρ. Α, ωραία. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους του Λαϊκού Κόμματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 75. Αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79. Αρχικό κείμενο ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 32 των φιλελευθέρων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 80. Αρχικό κείμενο ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 81. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 82 ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 84 του αρχικού κειμένου ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 85 του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Πρώτο, ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, πάλι ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό το τμήμα. Τροπολογία υπαριθμών 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαρίστως να επαληθεύσουμε, ήταν κάπως ε, κοντά το αποτέλεσμα. Επαληθεύουμε λοιπόν το 34. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Όντως, όντως εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται σαφώς. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κείμενο, ε, συγγνώμη, το κείμενο της αρχικής 90 σε τρία τμήματα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 95. Αρχικό κείμενο ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 96. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία υπαριθμών 20 σοσιαλδημοκρατών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 99 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 100. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο προβλέπεται ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Και αυτό το τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 48 της ομάδας ENF. Ε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται αυτή. Το αρχικό κείμενο της 101 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό το τμήμα. Τρίτο τμήμα πάλι ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 102. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται παρήθευση. Λυπούμε. Λοιπόν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 Δεύτερο, ονομαστική, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Γνωρίζω ότι είναι κοπιαστική αυτή η ψηφοφορία. Παρακαλώ σηκώστε όμως καλά τα χέρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Χρειάζεται επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία υπαριθμών 35. Πέρας. Σαφής έγκριση. Αλλά δυστυχώς δυσδιάκριτα. 119 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 120, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρο... Μπορούμε να επαληθεύσουμε εφόσον το επιθυμείτε. 36 ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία υπαριθμών 36. Πέρας. Απερίφθη. Υπαριθμών, αλλά τροπολογία λοιπόν, υπαριθμών 7. Ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο του εκτιμώντας δέλτα, ονομαστικά, αρχίζει. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, αιτιολογική σκέψη ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τρίτο τμήμα πάλι ονομαστικά αρχίζει πέρας εγκρίνεται και αυτό το τμήμα το G αρχικό κείμενο αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται το τμήμα αυτό, αιτιολογική σκέψη ήτα, η age, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, πέρας εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην ψηφοφορία επί του ψηφίσματος στο σύνολό του, ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος. Συγχαρητήρια στους συντάκτες του. Διακοπή τη συνεδρία.